Dear colleagues, good Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Να σας παρακαλέσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Επίσης, πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 8-12 Δεκεμβρίου και 16 Ιανουαρίου, εάν δεν έχετε παρατηρήσεις. Θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Ευχαριστώ. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτη, να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στις 5.30 το απόγευμα έχουμε κοινή συνεδρίαση βάσει του άρθρου 55 με τους συναδέλφους της Επιτροπής Γιούρη. για την ε, αποκάλυψη στατιστικών φορολογικών στοιχείων ε, για ορισμένες επιχειρήσεις και βάση της υποβολής έκθεσης αναχώρα και της σχετικής διαδικασίας. Όπως θα έχετε μάθει από τη Γραμματεία, αύριο στις 8 το πρωί θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με τη ΛΥΜΠΕ για να ψηφίσουμε για την πρόληψη Τη εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματο για σκοπού λεύκανση παράνομων προσόδων. Θα λάβουμε την απαραίτητη μέρημνα για τη διοργάνωση και των δύο συνεδριάσεων. Ε, Στι 16 Φεβρουαρίου είχαμε συνεδρίαση των συντονιστών και αυτό είναι η ανακεφαλαίωση των αποφάσεων, έλεγχος των κατεξόδου τη πράξεων. Στι 27 Μαρτίου θα επικεντρωθούμε στο PSD2 οι συντονιστές συμφώνησαν να οργανωθεί ανταλλαγή απόψεων στις 9 Μαρτίου στις 5 με τους ομολόγους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΖΑΣ για την οικονομική διακυβέρνηση, τον οικονομικό διάλογο και την ανταλλαγή με, τη, με τον πρόεδρο του Eurogroup. Θα έχουμε έκτακτη συνεδρία στις 21 Μαρτίου, τη ε, συνεδρία της Επιτροπής μας, στις 3 το απόγευμα. Επιτροπή έχουν θα ζητήσει να γίνουν δύο αποστολές στην Αθήνα και τη Λισαβόνα στα πλαίσια του, ε, των μακροοικονομικών ελέγχων στη CCCTB τώρα. Έχουμε αποφασίσει να καλέσουμε προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για να συμμετάσχουν σε μια από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας που θα εξετάσει το θέμα του CCCTB. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 αυτά. Τέλος, όπως θα γνωρίζετε, η Επιτροπή ΕΚΟΝ χωρίς πρώτο αντιπρόεδρο βρίσκει τον εαυτό της σε μια κατάσταση σχετικά ε, ασυνήθιστη. Το Προεδρείο της Επιτροπής δεν λειτουργεί επαρκώς, οπότε με τις παρούσες συνθήκες οι συντονιστές και εγώ αποφασίσαμε να απευθύνουμε έκκληση του αρχηγού των πολιτικών ομάδων για να βρούμε μια λύση στο δυνατόν συντομότερα και να μπορέσουμε να ε, συμπληρώσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής βάσει των κανόνων λειτουργίας που προβλέπει ο ιστορικό κανονισμό. Θα φροντίσουμε να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η διαδικασία και σε κάθε περίπτωση είμαστε πρόθυμοι να δράσουμε βάσει του εσωτερικού κανονισμού για να συμπληρωθούν όλε οι θέσει στο Προεδρείο. Έχετε κάποια παρατήρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς διερωτώμην. Έχουμε την ε, τελική προθεσμία. Ναι. Εκτός μικροφώνου. Ναι, με τις πολιτικές ομάδες. Είπαμε ότι αυτά περιμένουμε να γίνουν εν ευθέτω χρόνο. Δεν ε, θεωρώ απαραίτητο να σας πω την ημερομηνία τώρα, εδώ. Διαθεσμική διάλογοι, τριμερείς διάλογοι. Είχαμε στις 4 Φεβρουαρίου μια συζήτηση για την ε, καλύτερη χρηματοδότηση και το Finance Watch 2017-2020. Φτάσαμε σε πολιτική συμφωνία. Και αναμένουμε μετά τις τεχνικές συνεννοήσεις να ξαναρχίσουν ε, οι διαπραγματεύσεις στις 22 Μαρτίου 2017. και θα γίνει και άλλο τριμερή διάλογος για την ΕΦΡΑΚ. Τώρα επιτέλους μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5. Σημείο 5. Η εξέταση των τροπολογιών για τα ευρωπαϊκά νομία κινδύνου και τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά ταμεία. Η κυρία Πίτη Κάινεν, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν πολύπλοκα ζητήματα πολλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την έκθεση. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφωνία και απόκληση απόψεων και από των ε, γενικότερων ζητημάτων. Άρα σε όλα τα κεφάλια υπάρχει προθυμία να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τα με επιχειρηματικού κινδύνου. Εκεί που βλέπουμε βέβαια κάποια απόκληση απόψεων είναι πρώτον σε ό,τι αφορά τις κατώτατες επενδύσεις που απαιτούνται. Εδώ φαίνεται να υπάρχει υποστήριξη να μην πειράξουμε αυτό το κεφάλαιο το οποίο υπήρχε, είχε τεθεί στην αρχή. Ε, είχε γίνει βέβαια μεγάλη συζήτηση στην αρχή για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και το σχετικό κατώτατο όριο. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι χαμηλότερο το κατώτατο επενδυτικό όριο για ελληνικούς επενδυτές. Και όχι μια οροφή. Στο τεφάζ επενδύσεις. Για ποιο λόγο. Διότι σήμερα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ανάγκη για δανειοδοσία, αλλά υπάρχουν πολλοί ρηψοκίνδυνοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Όταν λοιπόν θέλουμε να ρυθμίσουμε τι επενδυτικέ ε, δυνατότητε ε, για του Ισλαμικού επενδυτέ, για να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα θέλουν υψηλή απόδοση με υψηλότερο κίνδυνο. Χωρί να σημαίνει ότι είναι και κερδοσκόποι. Υπάρχουν όμως κάποια πολύπλοκα ζητήματα, προϊόντα και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς που έγκυται ο κίνδυνος. Είναι υψηλότερη κίνδυνη στα τα επιχειρηματικού κινδύνου. Η ανανεώσιμη ε, ενέργεια, μια επένδυση, θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, ή το ένα ή το άλλο. Εγώ θεωρώ ότι καλό θα ήταν να γίνει δεχτή συμβαστική πρόταση. Δηλαδή, να δει η Κομισιόν τουλάχιστον για το μέλλον αν μπορούμε να έχουμε αυτή τη διαφορετική δομή για τους λιανικούς επενδυτές με ένα χαμηλότερο κατώτατο επενδυτικό όριο και ίσως να υπάρχει και μια οροφή βέβαια ταυτόχρονα των μέγιστων επενδύσεων για τους επενδυτές αυτού του είδους. Κατά τα λοιπά θα συμφωνήσω και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το με δυτικό όριο υπάρχει συμφωνία να μην το αλλάξουμε. Υπάρχει τώρα ε, ένα άλλο θέμα που είναι απαιτήσει δύο κεφαλαίων. Εδώ υπάρχει αρκετά μεγάλη ποικιλία απόψεων, από 100.000 και ένα τέταρτο των παγίων και κάποια άλλα. Αυτή είναι η πρώτη. Και απ' την άλλη υπάρχουν ε, άλλοι που λένε να μην υπάρχει καμία απέτηση για ίδια κεφάλαια και να είναι ένα ογδό του, των παγίων εξόδων τα ίδια κεφάλαια, όχι ένα τέταρτο. Εγώ προσπάθησα να αναζητήσω μια κοινή συνεννόηση για να προχωρήσουμε αργά όλοι μαζί σε ό,τι αφορά αυτές τις απαιτήσει, διότι γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Εμείς έχουμε τα διασυνοριακά ζητήματα, έχουμε τα μικρά ταμεία και όσο υψηλότερε είναι οι απαιτήσει, τόσο πιο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν νέα ταμεία και εκείνη το πρόβλημα. Γιατί χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, επιχειρηματικού κινδύνου ή σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Υπάρχει και άλλη πράγμα που λέει όμως. Τι γίνεται αν υπάρξει μια αποτυχία στο επιχειρηματικό κεφάλαιο, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Το να είναι 100.000 ή το 1 τέταρτο, το παγίο κτλ. δεν βοηθάει σε τίποτα. Άμα χάσει το 80%. Γιατί χάνουν όλοι. Λόγω της φύσης των επενδύσεων όλα αυτά. Γι' αυτό και είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. σε σχέση με του ελληνικού επενδυτέ. Βέβαια, οι επαγγελματίε ξέρουν περί τίνο πρόκειται και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τη θεμητή ανάγκη οι διαχειριστές των κεφαλαίων να ενεργούν υπεύθυνα, με υπευθυνότητα, νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με το άλλο θέμα. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εποπτεία, καταχώρηση και εποπτεία γενικά της δράσης ε, του Ταμείου. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Αφενός. Αφετέρου όμως, στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών, πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικά μια γνήσια αγορά πιερματικών κεφαλαίων. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, γιατί είναι διαφορετικοί οι κανόνες ανάλογα με το κράτος μέλος άλλα ποσά απαιτούνται για την εποπτεία, αλλιώς ερμηνεύονται οι κανονισμοί και αυτό βέβαια κάνει ιδιαίτερα δαπανηρό και δύσκολο για τα ταμεία να μπορέσουν να έχουν δραστηριότητα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Η αρχική μου πρόταση λοιπόν ήταν η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, να αναλάβει την καταχώρηση και όχι μια εθνική αρμόδια αρχή και να αναλάβει και την εποπτεία. Βέβαια, Πολλοί λένε ότι αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ίσως το Συμβούλιο να μην έχει την ιδιαίτερη πολιτική βούληση να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αφού λοιπόν συζητήσαμε με διάφορες πηγές και με την ΕΣΜΑ, καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση που προτείνω με τις τροπολογίες μου και που νομίζω ότι θα υποστηριχθεί από ορισμένες άλλες ακόμη πολιτικές ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν να έχει η ΕΣΜΑ ισχυρό ρόλο για να εξασφαλίσει την εναρμονισμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την εποπτεία, τη δεσμευριακή διαχείριση, τον ταμείο κεφαλαίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι αρμόδιες εθνικές αρχές τελικά θα επιφορτιστούν με την καταχώρηση και την καθημερινή εποπτεία. Η ΕΣΜΑ όμως θα έχει τη δυνατότητα και θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε καθοδήγηση και να ορίζει κοινά πρότυπα και κανόνες ό,τι αφορά την επικοινωνία, την εφαρμογή, την καταχώρηση, τις κατώτατες απαιτήσει, ε, εποπτεία κτλ. Και η ΕΣΜΑ επίσης θα έχει πλήρη πρόσβαση στα σφακέλους καταχώρησης και θα μπορεί να ε, επανεξετάζει τις διαδικασίες καταχώρησης ε, σε τακτά διαστήματα. Θα μπορεί επίσης να παρεμβαίνει σε επίπεδο μάλλον σε περίπτωση που είναι σαφές ότι η διαδικασία καταχώρησης δεν ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες ή δεν υπάρχει εποπτεία. Έτσι συνενώνουμε, αν θέλετε, το καλύτερο και των δύο διαφορετικών αυτών κόσμων. Και πιστεύω θα υπάρξει συνεννόηση και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ένα τελευταίο θέμα, εξίσου σημαντικό, είναι αυτό το διαβατήριο εμπορικής πρόθεσης ε, διαχείρισης. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά, αυτές οι ιδέες για αυτά τα δύο διαβατήρια. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε διαβατήριο και εμπορικής πρόθεσης και διαχείρισης. Αλλά αν δεν συμφωνούμε, ελπίζω τουλάχιστον η Κομισιό να το εξετάσει το θέμα και να προβεί σε κάποιες διευκρινήσεις ώστε να περιλαμβάνεται το διαβατήριο διαχείριση στα επόμενα βήματα, στα επόμενα στάδια της αναθεώρησης. Γιατί είναι αναγκαίο, ε, θα προσπαθήσω να προχωρήσω με το θέμα αυτό ώστε να τον πιο γρήγορα και βέβαια ο στόχος μου είναι να υπάρξει ένας στον δυνατόν ευρύτερος ε, συμβιβασμός για να είμαστε ενωμένοι ως κοινοβούλιο όταν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες εκ μέρου του κυρίου Κοτσολίνου, ο κύριος Μόργανο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Κοτσολίνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ για λόγους προσωπικούς και θα ήθελε να αναφέρω εγώ τα επιχειρηματά του στους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα τα διαβάσω όσο πιο καθαρά μπορώ. Καταρχάς, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και όλος ιδιαιτέρως την ε, συνάδελφο Πιετικάινεν. Σημειώνω θετικά διακείμενος ότι υπάρχουν πολλοί άριθμες τροπολογίες οι οποίες συμμερίζονται τις ανησυχίες και τις προτεραιότητές μου ακόμη και από βουλευτέ από διαφορετικέ χώρε και ασχέτω ε, πολιτική παράταξη. Άρα πιστεύει ο κ. Κοτσολίνο ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να βρεθούν συμβαστικέ λύσει με σημεία εφετερία τα εξή. Πρώτον, μια ανησυχία, το management passport. Υπό αυτή την έννοια, το επιτρέψουμε απλώ την ε, καταγραφή στο IMFD και το ESF την ε, διευκόλυνση του management διαβατηρίου δεν θα αλλάξει τίποτα, καθότι οι φορείς ε, Εδώ οι φορείς αυτοί δεν θα, δεν θα έχουν καμία ε, διευκόλυνση στη λειτουργία τους με το διαβατήριο διαχείρισης. Ε, η πρόταση της Επιτροπής λέει ότι η ΕΣΜΑ θα μπορεί να ορίσει το επίπεδο. Ο κ. Κοτσολίνο θεωρεί ότι το επίπεδο αυτό πρέπει να προβλέπεται από τον κανονισμό και όχι από το RTS μέχρι να βρεθεί το σωστό, ε, ο σωστός κανόνας και να υπάρχει βεβαιότητα δικαίου. Όπως και άλλοι βουλευτές, θεωρώ ότι πρέπει να υποβληθούν σχετικές τροπολογίες για τα δύο αυτά σημεία και επειδή υπάρχει περιθώριο για να επιτευχθούν συμβαστικές λύσεις, διατηρώντας την γενική δομή του κειμένου. Ως ε, τρίτο σημείο, η διάσταση των επιτροπών. Βάσει τη πρόταση τη Επιτροπή, η υποπτική Αρχή δεν μπορεί να υποβάλει ε, όρου στο κράτο μέλο υποδοχή. Ωστόσο, η λειτουργία εποπτεία και ελέγχου θα πρέπει να αναλαμβάνονται από τα ίδια αυτά τα ταμεία και να καλύπτονται και τα κόστη λειτουργία του. Και μάλιστα θα πρέπει να διαβαίνεται το πεδίο ε, αρμοδιότητα και κάποιε αρμοδιότητε ε, εποπτεία να, να, να τίθενται και στι ε, αρμόδιε αρχέ και να μην υπάρχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους εθνικούς φορείς οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν προμήθειες. Υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προμηθειών που να το καλύπτει η ίδια η πρόταση. Εν τέλει θα πρέπει να προβλέψουμε και περιθώριο για να σχολιάσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, την περιβαλλοντική μετάβαση δηλαδή. Τα κεφάλαια κινδύνου και της επιχειρηματικότητας μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά για να επικεντρωθούμε σε κάποιους περιβαλλοντικούς στόχους με περιβαλλοντικές ε, μεταβάσεις μέσω με την περιβαλλοντική μετάβαση που προβλέπει και το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Γιουρίκα. Οι διάφοροι φορείς και οι επιχειρηματίε θα πρέπει να ασχολούνται και με τι πραγματικέ συνέπειε των δράσεών του, των πρωτοβουλειών του. Ω εισηγητή λοιπόν Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα υποβάλει και τροπολογίε για να βελτιωθούν κάποια σημεία, όπω ε, και ο ισχυρότερο ρόλο τη ΕΣΜΑ. Άλλωστε υπάρχουν και τροπολογίε από άλλου συναδέλφου άλλων πολιτικών παρατάξεων που θα, ε, που θα κατευθυνθούν στον ίδιο στόχο, όπως με το διαβατήριο διαχείρισης. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθούν λύσεις εφόσον ενδιαφέρον από κοινού το ίδιο ε, ασχέτως της πολιτικής προέλευσης των βουλευτών. Ευχαριστούμε. επόμενο συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές, όχι. Γκουε, δεν βλέπω κανένα, ο κύριος Ούρτασον για τους πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ο δικός μας ο σχεδόν Λίπη, ο Φίλιπ Λαμπέρτς εξ ονοματός του να πω ότι θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτή τουλάχιστον τη φιλοδοξία εξέφρασαν όλα τα μέρη πριν από δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρθω σε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις του Φιλίπ. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε με την πρόταση της ηγήτριας να υπάρξει ένα καθεστώς το οποίο θα υποστηρίζει ένα διαβατήριο και εμπορίας ε, και διαχείρισης και συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει να κατέβει το κατόφλι για να επενδύει κανείς σε τέτοια ταμεία. Εάν τελικά συμφωνήσει και η πλειοψηφία θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν αναλόγως τα μέτρα προστασίας των λιανικών επενδυτών ε, σε ταμεία Ιούσεφ. Ε, επίσης, σημειώνουμε το ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες αυτή τη στιγμή προτείνουν απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων που αφορούν μόνο επιχειρησιακή συνέχεια με ένα επίπεδο που ανταποκρίνεται μόνο σε συνέχεια ολίγων εβδομάδων. Θεωρούμε όμως ότι οι απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων πρέπει να καλύπτουν και κάποιες ε, αναπάντεχες ε, ρευστοποιήσεις. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ποσοστό των κεφαλαίων υποδιαχείριση που θα μπορούσε να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του Ταμείου ή την ύπαρξη συμβατικών περιορισμών στην εξαργύρωση. Θα θέλαμε να επιμείνουμε στην ανάγκη να υπάρξει μια πιο προσεκτική προσέγγιση όταν μιλάμε για το ποια ακριβώς είναι τα επιλέξιμα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να αυστηροποιηθούν. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι θα πρέπει οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να ποικίλουν ανάλογα με τον χρονισμό της επένδυσης ε, κατά τη στιγμή της πρώτης επένδυσης θα πρέπει να περιορίζεται σε επιχειρήσεις ε, που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και με τζίρο κάτω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Στην δεύτερη επένδυση από την ΙΟΥΒΙΚΑ θα πρέπει να επεκταθεί σε επιχειρήσεις που ασχολούν μέχρι 499 άτομα και μέχρι τζίρο 50 εκατομμύρια και μετά σε όλες τις φάσεις των επενδύσεων δεν θα πρέπει όμως να υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει εμπορία σε μη ρυθμιζόμενες αγορές. Βεβαίως βλέπουμε ιδιαίτερα πως τα ταμεία αυτά θα πρέπει να παρέχουν στην ετήσια έκθεσή τους μια περιγραφή πρώτα απ' όλα το πώς, του πώς οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν την προσέγγιση τους και δεύτερον πώς ε, συνεισφέρουν στην καινοτομία οι επενδύσεις τους ε, με βάση τον πίνακα βαθμολογίας που έχει αναπτύξει η ΕΣΜΑ. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αξιολογεί και τον αντίκτυπο ex post στους στόχους Ένωσης. Uh, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω από άλλες πολιτικές ομάδες να ζητά κανείς το λόγο. Να ακούσουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο πρότεινε εδώ είσαι σχετικά είναι να μπορούμε να το στηρίξουμε. Θεωρώ πως η συγγήτρια έχει κάνει νομίζω μια πολύ καλή προσέγγιση για τη ρύθμιση αυτή. Η αναθεώρηση αυτής της ρύθμισης απαιτείται γιατί και οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχουν συνεισφέρει στον στόχο μας προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εξακολουθούμε να έχουμε πολύ περιορισμένες τέτοιες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ε, μετοχικού κεφαλαίου και βεβαίως παραμένουν τα ευρωπαϊκά ε, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου πολύ πίσω από τα άλλα διεθνή. Και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε μόνο εάν υπάρξει ένα διαβατήριο διαχείρισης το οποίο θα λειτουργεί στην πράξη. Και δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εστιάσουμε τόσο πολύ εκεί. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναλογική διαμόρφωση αυτού του διαβατηρίου γιατί τελικά θέλουμε να προωθήσουμε μια ε, ενιαία ευρωπαϊκή ε, κεφάλαια αγορά και όχι να έχουμε ένα μοσαϊκό. Επίσης η προστασία στην οδηγία δεν είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε. Υπάρχει λοιπόν το απαραίτητο ring fencing, αλλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι κάτι το συγκρίσιμο με άλλες ε, καταστάσεις βεβαίως. Αυτό εξαρτάται και από την ε, τάξη μεγέθους, οπότε έχει δίκιο η ΣΕΠΑ όσον αφορά τις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια αρεαλιστική προσέγγιση το να δώσουμε αρμοδιότητες στις, ε, στην ΕΣΜΑ, την οποία δεν ζήτησε καν και δεν ξέρουμε αν μπορεί και να τις εκπληρώσει, δεν νομίζω να είναι πάρα πολύ σωστό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Περβάμος Μπερές. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πνεύμα με τον οποίο επεξεργάζεται την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Πράγματι ήταν κοινός ο στόχος και η νομοθεσία που επεξεργαστήκαμε από ό,τι φαίνεται δεν επιτυγχάνει τον κοινό Άρα, αναμφίβολα είναι ώρα να κάνουμε μια αναθεώρηση της κατάστασης. Πολλές παρεμβάσεις αναφέρθηκαν στο ρόλο της ΕΣΜΑ. Νομίζω ότι εξορισμού σε μια τέτοιου είδους νομοθεσία πρέπει να εμπιστευτούμε τις δομές που έχουμε δημιουργήσει, όπως την ΕΣΜΑ δηλαδή, ώστε η νομοθεσία να είναι ευρωπαϊκή και προοδευτική. Νομίζω ότι η ευκαιρία αυτής της αναθεώρησης θα πρέπει να ενδιαφερθούμε για τα συμφέροντα και των ιδιωτών ε, επενδυτών και για το legal entity identifier εγώ ζητώ να προσδιοριστεί ιδίως αν θέλουμε ενιαίους κανόνες και προσέγγιση ο κ. Κοτσολίνο είναι ο σκιώδης ηγητής, ακούσαμε να λέει τις απόψεις του κ. Μόργανο. Μίλησε και για τις προμήθειες, να μην επιβάλλονται προμήθειες και σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τα άλλα κράτη να προβαίνουν σε εποπτεία αλλά την προσπάθεια που αυτό συνεπάγεται να μην τη λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική εποπτεία, αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και έρχομαι στα πιο λεπτά, ίσως το πιο λεπτό ε, σήμερα. Το level playing field θα το έλεγε ένας φρυξελιώτης. Μεταξύ αυτών των δύο ταμείων εταιριών. Έχουμε το ζήτημα του διαβατηρίου. Αν θα εκδίδεται υπό τις ίδιες ε, συνθήκες, υπό τους ίδιους όρους, ναι ή όχι. Και τι θα απαιτούμε, ποιες θα είναι οι απαιτήσει από τα ταμίκνυμα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με αυτό που απαιτούμε στο πλαίσιο TFMD. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την εποπτεία αυτών των ταμείων και εταιριών. Θέλουμε να αυξήσουμε την ελκυστικότητά τους, δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε και νέα hedge funds στο όνομα της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της χρήση των κεφαλαίων. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι κάνουμε μια λάθος επιλογή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλο τον λόγο. Θα ακούσουμε τώρα τον πρόσφατο της Κομισιόν, τον κύριο Γκέπνερ. Να Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Να σας υπενθυμίσω. Και συμφωνώ με την αξιολόγηση που έγινε πριν. Από όταν το 2013 είχαμε τα δύο αυτά πλαίσια, είχαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά όχι ίσως αρκετή επιτυχία. Γι' αυτό επανερχόμαστε με την αναθεώρηση τόσο σύντομα. Όταν μιλάμε στον κλάδο και στην διαβούλευση και στην στοχευμένη διαβούλευση που έγινε ήταν σαφές ότι μας είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα υπήρχαν κάποιοι κλάδοι και κατά την άποψη του κλάδου όπου κάποιες βελτιώσεις θα βοηθούσαν το να γίνουν τα πλαίσια αυτά πιο επιτυχή. Να σας δώσω ένα νούμερο. Είμαστε πίσω από τις ΙΠΑ όσον αφορά το μέγεθος ε, των αγορών αυτών ε, και όσον αφορά τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύου αλλά και το σύνολο της αγοράς οπότε θεωρούν πως υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι δύο βασικές αλλαγές ε, που προτείναμε είναι πρώτα απ' όλα να ανοίξει η διαχείριση σε μεγαλύτερους διαχειριστές και χαίρομαι για το ότι οι περισσότεροι συνεισηγητές σήμερα συμφωνούν. Θεωρούμε ότι έτσι θα υπάρξει δυνατότητα εμπορίας σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο επενδυτών και σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές και τελικά θα βοηθήσει και τη Σίγιου και τη Γιούσεφ να είναι κάτι το έμπιστο και να φτάσουν σε πολύ περισσότερους επενδυτές. Το δεύτερο θέμα για μας είναι βεβαίως ο ορισμός ε, των επιλέξιμων στοιχείων ε, ενεργητικού. Θεωρούμε ότι έτσι και τα δύο πλαίσια θα γίνουν πιο ελκυστικά. Θα υπάρξει η δυνατότητα μιας ε, μεγαλύτερης διασποράς του κάθε χαρτοφυλακίου. Και βεβαίως ακολουθώντας την λογική ότι ο στόχος είναι να γίνει το πλαίσιο πιο ελκυστικό, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει νόημα να πειράξουμε το όριο των 100.000 ε, για, ε, ε, για το κατόφλι. Κανείς δεν θεωρούσε ότι υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό. Επίσης, η απέτηση αυτή των 100.000, το εισιτήριο το λεγόμενο, ε, θεωρήθηκε ένα πάρα πολύ απλό ε, τεστ, ενώ τα υπόλοιπα τεστ της ΕΛΤΙΦ τα θεώρησε ο κλάδος ε, κάπως πιο περίπλοκα. Δηλαδή το να μιλήσουμε για την γενικότερη οικονομική κατάσταση των επενδυτών. Οπότε αυτό πρέπει να το κρατήσουμε γιατί λειτουργεί. Για την απέτηση των ιδίων κεφαλαίων. Για εμάς ε, και πάλι ο στόχος είναι τα δύο αυτά πλαίσια να είναι ελκυστικά για τους ε, διαχειριστές ε, να μπορούν εύκολα να στηθούν και δεδομένου του ότι υπάρχει ήδη κάποια εγγύηση θεωρούμε ότι η απέτηση των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι πολύ πιο ελαφριά σε σχέση με το IMFD. Η αρχική μας πρόταση ήταν να αφήσουμε να το διαχειριστεί αυτό η ΕΣΜΑ, αλλά οποιαδήποτε λύση επιτυγχάνει τους στόχους αυτούς ε, θα μας ικανοποιήσει και αυτό σημαίνει βεβαίως ένα πιο ελαφρύ ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι απαιτήσει αυτές βεβαίως επιβάλλονται στην εταιρεία διαχείρισης, όχι στο ταμείο, ούτε στους επενδυτές εάν πάει κάτι στραβά. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο να αποσμειώσει του επενδυτέ αν πάει κάτι στραβά. Αυτό είναι άλλη υπόθεση και έχουμε άλλα μέσα γι' αυτό. Για το θέμα του διαβατηρίου της διαχείρισης, το λεγόμενο, δεν βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη απέτηση από μικρούς διαχειριστές να φτιάξουν κάτι εκτός του κράτου μέλους τους. Οι μεγαλύτεροι ή άλλως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριο ανησυχούμε ότι εάν τώρα ε, φτιάξουμε ένα τέτοιο πλαίσιο θα αφορά αρκετές αλλαγές στο κείμενο και θα καθυστερήσει την όλη διαδικασία και ανησυχούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι χειρότερο από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Να καταλήξουμε με πιο πολύπλοκη κατάσταση και πολλούς και διαφορετικούς κανόνες ε, για το ποια είναι η χώρα προέλευσης ε, και κατάληξης και βεβαίως θα πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα όταν θα μεταρρυθμίσουμε την FMD, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να ανοίξουμε το θέμα. Επίσης, σημειώνουμε τις προτάσεις σας για έναν πιο έντονο ρόλο της ΕΣΜΑ. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή προετοιμάζει μία αναθεώρηση και χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ε, το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορούμε ε, να σας δώσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο ως πληροφορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και τώρα πάλι η Συγήτρια. Θα ευχαριστήσω τους Κιώδης και την Επιτροπή για τα σχόλιά τους. Thank you. Ευχαριστούμε. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 22 και 23 Μαρτίου. Και μετά θα αρχίσουν οι τριμερείς διάλογοι. Ωραία. Κλείνουμε με το σημείο αυτό. Και περνάμε στο σημείο 7. Γιατί το 6 μετακινήθηκε στο αυριανή συνεδρίαση. Και τώρα, το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017 και παράταση 2018-2020. Δισεκητής είμαι εγώ ίδιος, ο πρόεδρός σας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αδρές γραμμές της έκθεσής μου ούτως ή άλλως, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες ε, των τροπολογιών, έχω εντοπίσει κάποιους, κάποια πεδία όπου οι, δεκεντρώνονται οι, τα σχόλια των συναδέλφων. Πρώτη ομάδα τροπολογιών, η ανάπτυξη συνολικών δικτών για την κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων στην Ένωση. Άλλη, ανάπτυξη μεθοδολογίας για την μελέτη που εξετάζει την ισότητα των φύλων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επίσης, δείκτες για την απασχόληση με διάκριση μεταξύ απασχόλησης μερικού ή ε, πλήρους χρόνου, των σταθερών ή ε, των ε, μερικού χρόνου συμβάσεων και την ποιότητα της απασχόλησης. Επίσης, το τι γίνεται στην περίπτωση ενδεχόμενης αποχώρησης κράτους μέλους από την Ένωση. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα των τροπολογιών. Νομίζω ότι όλες είναι λογικές, μπορώ να τις συμμεριστώ και τις περισσότερες να τις δεκτώ. Δεύτερο πεδίο για τους δείκτες του ΑΕΠ και τους σχετικούς ε, δείκτες, το βιωτικό επίπεδο, την ποιότητα ζωής, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τις εξωτερικές συνέπειες από την σκοπιά πάντοτε των εθνικών λογαριασμών. Τρίτον, πολλές τροπολογίες υποβλήθηκαν για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ε, συναθρισμένων δικτών για την ποιότητα του εισοδήματος και τέλος τροπολογίες που ζητούν πρόσθετη υποβολή στοιχείων για τα στατιστικά προγράμματα των Εθνικών Φορέων των και για την πρόοδο της χρηματοδότησης των ε, παραμέτρων που κάνουν τις στατιστικές πιο φιλικές προς τους χρήστες, όπως τη διάθεσή του στον ιστότοπο και την διαθεσιμότητά τους στην ευκολία πρόσβασης. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους και τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις συμβαστικές λύσεις. Μέχρι να καταλήξουμε, ελπίζω εύκολα, σε συμβαστικέ ε, τελικές λύσεις. Ευχαριστώ. Σκιώδης από το ΕΛΚΟ, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου για το έργο να σα συγχαρώ όλου. Όπω είπατε, οι τροπολογίε πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Το έγγραφο, ο κανονισμό ε, δεν ε, υφίσταται και κάποια ουσιαστική αλλαγή. Έχει βάλει στις 10 προτεραιότητες της Κομισιόν την ανάγκη ε, για την κάλυψη της ζήτησης στατιστικών στοιχείων. Και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του εγγράφου. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής ε, Ένωση θα πρέπει να βασίζονται ακριβώς ε, σε μια στατιστική πληροφόρηση υψηλού ποιότητας. Τα συγκρίσιμα βέβαια ε, στατιστικά στοιχεία είναι κάτι σημαντικό και σε στατιστικό και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να υπάρχει μια αντίστοιχε απαιτήσει. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι τους τρεις βασικούς στόχους που τόσε φορές του έχουμε αναφέρει. Ε, έχουμε δηλαδή στατιστική πληροφόρηση υψηλή ποιότητα. να μπορούμε επίση να ανταποκριθούμε πολύ πιο γρήγορα στις ανάγκες της Ένωσης για τα στοιχεία και τρίτον να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι τους τρεις αυτούς στόχους με το έγγραφο αυτό τους ε, εκπληρώνουμε και δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από παρά ένα ακόμα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές δεν βλέπω να είναι κανείς. Ο, από τους φιλελεύθερους ο κύριος Χαμπών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, διότι νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν είναι αμφίμαχο, δεν, επιλεγω... δεν είναι επίμαχο. Και... Βλέπουμε για μια ακόμη φορά στην Ευρώπη ότι δεν έχουμε φιλόδοξο προπολογισμό και δεν έχουμε κάποια φιλοδοξία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εσείς αναφέρετε ορισμένα στοιχεία ως εισηγητής κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες για στατιστικά στοιχεία. Έχουμε πραγματικά γελία από εσάς στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τις καλύψουμε τις ανάγκες αυτές παρότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτήν την έννοια, η Άλντε πραγματικά ενδιαφέρεται τα μάλα για την ε, ενίσχυση ε, των δυνατοτήτων ανάλυσης του μεγάλου προβλήματος ανισοτήτων που έχουμε και της διεύρυνσης αυτού του χάσματος. Και δεν μιλάμε μόνο για το δίκτυ αλλά για πολλές άλλες ε, μετρήσεις και δείκτες που δεν φαίνονται να είναι χρήσιμοι δεν υπάρχει καλή κατανομή, ε, ισομερής κατανομή της ανάπτυξης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στο σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ο προλαλή σα είπε ότι πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστέ σε διεθνέ επίπεδο κτλ. Πέραν τη συγκυρία. Πρέπει να έχουμε σταθερά στατιστικά στοιχεία συν το χρόνο. Και όχι μόνο με βάση το τι αποφασίζει κατεπηγόντω ένα επίτροπο σήμερα. χάρη, μετανάστε σήμερα, ναι. Όχι, πρέπει να έχουμε ένα σημαντικό σώμα στατιστικών στοιχείων γενικά. Σταθερό. Επίση, για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Άμεσα πρέπει να καταρτίζονται μέσω μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ε, στατιστικών ε, στοιχείων, έστω και με μικρά βήματα. Είναι κάτι το καλοδεχούμενο. Ποια είναι η ανεργία στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία. Κάποιοι το λένε. Δεν ξέρω πόσους μπορεί να ενδιαφέρει. 5-10 χιλιάδες για την ανεργία στη Ρωσία. Βέβαια δεν θα δώσουν το σωστό στοιχείο, θα το δώσουν απλά στο στοιχείο, αλλά και τα λοιπά. Τώρα τα πάρουμε όλα και να τα βάλουμε μέσα σε ένα καλάθι χωρίς να έχουμε υπολογισμού. Τι να πω. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε η μεθοδολογία να είναι παρόμοια σε κάθε χώρα. Αν δεν έχουμε συγκρίσιμα εγκεκριμένα στοιχεία, ε, είναι χειρότερο και από αυτό που έλεγε ε, η Ισραηλινή ότι η, η στατιστική είναι ο πιο ε, κομψός τρόπος να λες ψέματα. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε με τα λίγα μέσα που έχουμε στα δεσί μας να βελτιωθεί στον το περισσότερο αυτό το στατιστικό σύστημα. Και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ανισότητες και να εστιάσουμε στην πραγματική δημοσιονομική ικανότητα δεν ξέρω αν γίνεται να ληφθούν υπόψη όλες οι υποδείξεις που κάνετε ή τέλος πάντων ε, να εστιάσουμε σε ένα-δυο πράγματα μόνο στην πρώτη φάση. Αυτά έχω να πω ε, εκ μέρους άλλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το έργο σας στο συγκεκριμένο φάκελο. Thank you. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κύριος Γκίγκολντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς σε ευχαριστώ για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που έχει διάφορα πράγματα που μας ενδιαφέρουν όπως δείκτες που αφορούν την έμφυλη βία, κοινωνικά στατιστικά στοιχεία, ζητήματα μετανάστευσης που πρέπει να καλύπτονται πολύ περισσότερο όπως και το ευρύτερο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Πέρα από αυτό, νομίζουμε ότι έχει φτάσει η ώρα να ξαναδούμε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα και να ξαναδούμε τη δουλειά που κάναμε πριν από λίγα χρόνια. Κάποια από τα πράγματα που είχαμε συντάξει με τον συνομοθέτη δεν έχουν εφαρμοστεί. Και είναι σημαντικό αυτό για τον διάλογο με την Eurostat και να δούμε το τι έχει εφαρμοστεί και το τι όχι. Οπότε προτείναμε κάποιες τροπολογίες για να επιθυμήσουμε κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και θα ήθελα να επαναλάβω κάποια από αυτά. Πρώτα απ' όλα οι δείκτες της Ευρώπης 2020 ε, είναι ακόμα ξεπερασμένοι και τα πιο πρόσφατα δεδομένα που έχουμε είναι του 2014. Οπότε, εάν είναι αυτή η βασική μας στρατηγική, θα πρέπει να έχουμε δείκτες πιο πρόσφατους από το 2014 κατόπιν. Το πόσο φιλικό είναι το site και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, δεν είναι στο ιδανικό σημείο. Έχουμε άλλα site στατιστικών υπηρεσιών που το καθιστούν πιο οικολόγια δασκάλους, για φοιτητέ να φτιάξουν διαγράμματα με τα δεδομένα, να κάνουν παρουσιάσεις για το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Μέχρι στιγμής ε, το site της Eurostat ε, χρειάζεται να κάνει κανείς εισαγωγή για το πώς χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία λογισμικού. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Ε, και είναι σημαντικό νομίζω αυτό για να έχει και μια προσθέμενη αξία για τον πολίτη. Και επίσης θα θέλαμε, όπως αποφασίσαμε και στο προηγούμενο πρόγραμμα, οι δραστηριότητες κοινωνικής οικονομίας να μετρούνται σαφώς όπως προτείνει ο ΟΗΕ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στην Ευρώπη. Οπότε κάναμε αρκετές προτάσεις. Επίσης, χαιρόμαστε για το ότι αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει σημαντικές προτάσεις όπως η Άλντε και οι Σοσιαλδημοκράτε για την ανισότητα, η Αριστερά για τη φοροδιαφυγή, το ΕΛΚ για ε, Ε, κάπως πιο εδαφική κατανομή των στοιχείων και ο κύριος Σώνας Φερνάνδης για την κυκλική οικονομία και η Νίνα Τζίλ για τους δείκτες απασχόλησης. Και όλα αυτά είναι χρήσιμες ιδέες και θα ήθελα να ακούσω από την Eurostat τι από όλα αυτά θα μπορούσε να εφαρμόσει και μέχρι πότε μπορούν να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόσουν ε, το παλαιό πρόγραμμα ε, στατιστικών στοιχείων. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο από τους και εισηγητές. Ούτε, ούτε κανέναν γενικός. Α, ναι, παρακαλώ. Και όσο κανεμάνες. Η κυρία Κάπελ ζητάει συγγνώμη γιατί και εκείνη απουσιάζει και έχει κάποιες παρατηρήσεις. και να σας πω εξής, ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία για να μετρήσουμε την πρόοδο των, ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θεωρεί ότι η λέξη πρόοδος είναι ένας όρος κανονιστικός ε, και θα πρέπει να μιλάμε για τα ευρήματα και όχι για πρόοδο των ε, πολιτικών της Ένωσης και μια δεύτερη παρατήρηση μιλάτε για νέες ε, προβολές πληθυσμού και την γύρανση και θα πρέπει να προσθεθεί και η δημοκρατική εξέλιξη με βάση τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια ποσοστά γέννησης, το κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη παρατήρηση, στατιστικά κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να προσέξουμε, θεωρούμε πάρα πολύ τα πρόσφατα γεγονότα και διαπιστώσεις ε, τα νούμερα αυτά και να αποφύγουμε να επιλέγουμε ή να επιλέγουν οι επιστήμονες μόνο όσα τους συμφέρουν. Τέταρτον, λέει εδώ πέρα assumes ε, ότι η Κομισιόν υποθέτει ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους του κανονισμού και πρέπει να γίνει αυτό στο επίπεδο της Ένωσης. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο στήριξη αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζει αλλά όχι να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη και να λέμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτερ Εβεράς, ο Γενικός Διευθυντής της Eurostat, είναι εδώ μαζί μας. Παρακαλώ σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και επειδή θα μιλήσω τελευταίο, να πω ότι είμαι διευθυντή τη Eurostat, υπεύθυνο για την ελληνική κυβέρνηση και νομικό πλαίσιο για τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ γενικώ. Πρώτα απ' όλα να, ευχαριστα... να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου προ τον ε, καθήλυνα αρμόδιο συγκεκριτή και του Σκιώδη και για όλα τα σχόλια και τι τροπολογίε που αποβλήθηκαν για το σχέδιο έκθεση. Το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή σα ανέκαθεν στήριζαν τις στατιστικές τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχουν συνολικότερα ευρωπαϊκά στοιχεία και να συνατρίζονται ε, να υπάρχει συμπίληση έγκαιρη. Η Επιτροπή σα πάντοτε στήριζε την Eurostat ώστε να υπάρχει μεγάλη ποιότητα στην ε, τροφοδότηση του συστήματος και την παραγωγή, ώστε να διευκολυνθούν ε, οι υπεύθυνοι των αποφάσεων και γενικώ οι πολιτικοί ηθήνοντες παρά τις ταραχώδεις τελευταίες περιόδους όπου η συγκέντρωση πληροφοριών μας ανάγκασε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικές μεθόδους, συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας. Το στατιστικό πρόγραμμα από το 2018 στο 2020 με την παράτασή του σημαίνει ότι δεν θα ανακαινήσουμε πλήρως ε, το πρόγραμμα, ούτε θα χρησιμοποιήσουμε εκ νέου πλήρω το πρόγραμμα του 2013-2017. Αλλά δεν θα αρχίσει και ένα τελείω νέο κύκλο. Η παράταση θέλει να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματο, ώστε να εκπληρώνει τα άλλο και υψηλότερα πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί και να καλύπτει τι υψηλέ απαιτήσει. Με του τωρινού πόρου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια όθηση για το μέλλον και να καλύψουμε ε, αρκετή δουλειά. Θα πρέπει να ενοποιηθεί το σύστημα, να εξορθολογιστεί και ταυτόχρονα να επιδιώξουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας βάσει των σημερινών πολιτικών αναγκών. Γι' αυτό, όπως θα προσέξετε στην πρόταση, πραγματικά έχουμε σκεφτεί κάποια βήματα που τεχνολογικώς έχουν αποδείξει την αξία τους ε, για να εξασφαλίσουμε ποιοτικά στοιχεία όπως για τη μετανάστευση, την κοινωνική ε, κινητικότητα και άλλα στοιχεία που αναφέρετε κι εσείς. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί σας ε, κατά λεπτό στη διάρκεια των επερχόμενων αντιπραγματεύσεων και άλλες ιδέες όπω την τροπολογία 23 για τα θέματα τη μετανάστευση, την 63 που είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, την 62 και 84 για την παρουσίαση στον ιστότοπο. Θα επανέλθουμε σε αυτό, αυτό που είπε ο κύριος Γκίγκολτ και μετά για την 35 ε, και 47 για την ενέργεια και την 48 που είναι για τη γεωργία. Ο διάλογος νομίζω μας επιτρέψει να περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λόγου χάρη, η τροπολογία 63 που προτείνει βελτίωση τη διαθεσιμότητα των δικτών για τον έλεγχο τη στρατηγικής 2020 για την επιδίωξη των στόχων. Το ανέφερε και ο κ. Γίγκολτ. Είμαι σχεδόν βεβαίω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι η έγκαιρη παραγωγή των δεδομένων είναι καθοριστική σημασία για την Eurostat. Όμω, όλοι επίση θα καταλαβαίνετε ότι ένα στοιχείο είναι να παράγονται έγκαιρα, ένα άλλο να είναι και ακριβή τα στατιστικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία για τον κάθε δείκτη ξεχωριστά, ώστε να βεβαιωθούμε ότι συνολικά υπάρχει ποιότητα. Διότι η υψηλή ποιότητα βεβαίω έχει άμεση συνάρτηση, είναι σε άμεση συνάρτηση με το έγκαιρον. Είναι πέντε οι θεματικές ενότητες της Ευρωπαϊκής της Στρατηγικής του 2020 και αυτό όπως ε, λέγεται πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πεντάμινο όπως ζητάει η τροπολογία 63. Μόνο σε ένα τομέα δεν συνέβη όμως αυτό τον τομέα των κλιματικών αλλαγών. Εκεί που τα πράγματα είναι λίγο πιο κειμενόμενα. Να το πω το γιατί. Κάποια από τα στοιχεία όπω η κατανάλωση τη ενέργεια βασίζονται σε ε, εθελούσια υποβολή των στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Πρέπει δηλαδή εκεί να επιτελεστεί πρόοδο. Δεν υπάρχει επίση ε, δεσμευτική ε, καταληκτική προθεσμία. Και μάλιστα τα δεδομένα ε, αποστέλλονται περίπου ένα δίμηνο μετά το, τη λήξη τη 12 ε, προθεσμία. Λόγου χάρη για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, αυτά αποστελούνται πολύ αργά και είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Βεβαίως, για τους δείκτες και το σύνολο των δικτών, ε, παρακολουθούμε τις απαιτήσει που υπάρχουν και την ζήτηση από την πλευρά των πολιτικών εθνόντων και θα προσπαθήσουμε στην, ε, στον εξοφυλλογισμό των διαδικασιών και τη δουλειά μας να τα ενσωματώσουμε. Επίσης για τη συνεχή επικαιροποίηση των επιγραμμικών λιμάτων για τους ε, στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του 2020. Μόλις ε, λαμβάνουμε τα δεδομένα φροντίζουμε να επικαιροποιούμε τον ιστότοπο. Έτσι μπορεί η ετήσια έκθεση για την ε, παρακολούθηση της επιδίωξης των στόχων του 2020 να είναι και πάντοτε σε συνάρτηση με τα στοιχεία για την 62 και 84 που αφορούν την παρουσίαση των στοιχείων στον ιστότοπο της Eurostat ε, περίμενα ε, σχόλια και τροπολογία και γι' αυτό, αλλά να πω ότι για την ε, Eurostat. Το να είναι φιλική προ το χρήστη στι σελίδε τη, στον ιστότοπό τη, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρώτη μα προτεραιότητα και στην πολιτική την, επικοινωνία, την επικοινωνιακή μα. Άρα, η φιλικότητα προ το χρήστη, η πιο εύκολη πρόσβαση για όλε τι ομάδε χρηστών στον ιστότοπο και η απλή παρουσίασή του είναι πολύ σημαντικό. Ο Eurostat έχει καταβάλει πολλέ προσπάθειε τα τελευταία χρόνια στην επικοινωνία των στατιστικών στοιχείων και στην βελτίωση του ηθοτόπου. Για παράδειγμα, εισάγοντα κάθε είδου διαδραστικέ απεικονίσει με χάρτε, διαγράμματα κ.ο.κ. Σε γενικέ γραμμέ, μάλλον τον Ιανουάριο, πριν από μια-δύο εβδομάδε μάλιστα, ε, ο ιδιότοπο μα ε, ανανεώθηκε πλήρω με την εισαγωγή ενό νέου συνόλου που καθημερινά ε, παρουσιάζει την δημοσίευση νέων εργαλείων, καθώ και το Twitter τη Eurostat, που είναι πολύ αποτελεσματικό ώστε να ενημερώνει του νέου χρήστε και έχει γίνει πολύ δημοφιλέ. Επίση, να πω ότι συστηματικά λαμβάνουμε θετικά σχόλια για τις πρόσφατες βελτιώσεις μας, λόγω χάρη από την κοινότητα των χρηστών, όπως εκπροσωπούνται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Στατιστικών. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίε σε εξέλιξη. Και είμαι και εγώ πεπισμένο, όπω και εσεί κύριε Γκίγκολτ, ότι υπάρχουν και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Όμω δεν έχουμε πάυσει να εργαζόμαστε με τη τροπολογία σα, θα βρούμε και άλλο πάτημα για να συνεχίσουμε να είμαστε εξίσου εργατικοί. Και βεβαίω θέλουμε ο στόχο τη Eurostat να είναι κάτι που θα τα ανταποκρίνεται στι προσδοκίε των πιστών και θα είναι στο επίπεδο άλλων ανάλογων στατιστικών ιστοτόπων. Περιμένουμε και την ε, μελέτη που θα δημοσιευτεί στο δεύτερο εξάμεινο τη Βρετανική χρονιά για να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Για τις άλλες τώρα θα μπορούσα να δώσω και άλλα σχόλια και να απαντήσω, να αντιδράσω, αλλά περιμένω Εδώ θα πει και ο συγκεκριτή για να προσθέσω ίσω περισσότερε παρατηρήσει. Απλώ να ολοκληρώσω λέγοντα λέγοντας ότι η πρόταση νομίζω πω στέλνει ένα σαφέ μήνυμα. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα πρέπει να ανταποκριθεί σε νέε απαιτήσει και προσδοκίε. Πραγματικά λοιπόν θέλουμε να υπάρχει μια καλή χρήση του προπολογισμού και τη ευρωπαϊκή στατιστική που θα φέρει σημαντικές, σημαντική προστιθέμενη αξία και θα βοηθά τα στατιστικά συστήματα των κρατών μελών. Παραμένουμε βέβαιοι ότι με τη δική σας στήριξη για μια μικρή αύξηση στα κονδύλια και χωρίς ιδιαίτερη αιρεσιμότητα στην ε, εκτέλεση των κονδυλίων αυτών από, τα, από τη Eurostat με τις, ε, με τις συνηθισμένες πρακτικές που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται ελπίζουμε ότι στις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές θα μπορέσει να ενταχθεί και αυτή η μικρή αύξηση. Και υπολογίζουμε στη δική σας στήριξη. Σας ευχαριστούμε κύριε Σεγητά και την Επιτροπή σας για τις προτάσεις σας και την ε, διαρκή σας στήριξη για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε στη διάθεσή σα για περισσότερε απαντήσει ή διευκρινήσει εφόσον χρειαστούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Also... Ευχαριστώ την Κομισιόν αλλά και τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω ότι έχουμε μια ευρύ κοινή βάση εργασίας. Η Στατιδά μου τη συμφωνεί με ένα μεγάλο μέρος ε, των παρατηρήσεων των συναδέλφων. Σε κάποια υπάρχουν διαφωνίες, αλλά εν γέννη είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε καλές συμβαστικέ προτάσεις για να μπορέσουμε βέβαια να υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τη σχετική νομοθεσία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο. σε σχέση με όσα είπα. Νομίζω ότι είναι λογικές προτάσεις που άκουσα. Απλά τώρα θέλουμε να τις επεξεργαστούμε, να βρούμε την ακριβή διατύπωση. Αλλά είμαι αισιόδοξο όπως είπα, για τη τελική έκβαση. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Εξέταση, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι. Όχι, λάθος. Α, 27 Μαρτίου, α, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι, 27 Μαρτίου ψηφίζουμε, ναι, ναι. Λέω και εγώ 27 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ την συνάντηση της Επιτροπής. Ακολουθεί μετά από ένα σύντομο διάλειμμα η κοινή συνεδρίασή μας